και Ένωση. Είναι η ετήσια έκθεση για το έτος 2015. Έχει την σκητάλη ο κύριος Γκουαρτιέρη για τέσσερα λεπτά. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η Τραπεζική Ένωση είναι το πιο σημαντικό βήμα, ούτως ώστε να έχουμε ε, μια αυθεντική νοσηματική ένωση από τότε που θεσπίστηκε το ευρώ. Να υπάρχει ενιαίος ευωτικός μηχανισμός και κάτι το οποίο θα είναι σημαντική μετά τη αρμοδίτητων από την Ευρωζώνη προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για μια σταθερότητα και ε, εμπιστοσύνη προς τις τράπεζες ούτως ώστε να κατανείμουμε τους κινδύνους γιατί έτσι θα αναβαθμίσουμε την ε, Τραπεζική Ένωση η ολοκλήρωση. Όμως αυτή η μεταφορά αρμοδιοτήτων θα ε, απαιτεί και κοινολογικό έλεγχο. Να και αυτή η έκθεση είναι η έκφραση αυτού του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σε σχέση με αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές μου για την συνεργασία, αλλά και τη γραμματεία και το επιτελείο μας για την εργασία τους. Επίσης ήταν ε, ο διάλογος ε, με ανοιχτό ε, πνεύμα και με διαφάνεια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ενιαίο υποπτικό μηχανισμό και οπότε πετύχαμε και από πλευράς λειτουργικής και από πλευράς ποιότητας της εποπτείας. Ταυτόχρονα δε όμως εντοπίσαμε κάποια προβλήματα, υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων και στην εποπτεία και στην εξυγίανση, δηλαδή τονίσαμε το πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική λειτουργία συντονισμού για τις ε, πολιτικές του μηχανισμού εξυγίανσης και επίσης χρειάζεται σταθεροποίηση του εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου. Επίσης πρέπει να βελτιώσουμε το ότι οι τράπεζες θα πρέχουν μια κοινή ε, προσέγγιση εποπτείας και αυτά τα microprudential μέσω της μικροπροληπτικής λειτουργίας τους. Χρειάζονται σαφήνεια, χρειάζονται ε, ξεκάθαρο τοπίο οι τράπεζε όσον αφορά τι ε, κεφαλικέ απαιτήσεις αλλά αυτό δεν ισχύει με το MDR γιατί λέει η έκθεση ότι εδώ δεν υπάρχει ξεκάθαρο τοπίο, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίσει το μηχανισμό να έχει την ευελιξία, ούτως ώστε να μην έχουμε κάποιες οίκιστα ευέλικτες λύσεις που να ε, έχουν κακέ επιπτώσει στην ε, αγορά των ομολόγων. Άρα θα πρέπει το MDA να ξεκαθαριστεί, αλλά επίσης και η λειτουργία του δευτέρου πυλώνα κάτι το οποίο αφορά συγκεκριμένου κινδύνου. Και αυτά τα είδαμε και χθε στο σημείο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχή η διαδικασία τη αναθεώρησης και θεωρούμε ότι ο SSM θα πρέπει να καλύψει πλήρω και να λάβει όλα αυτά υπόψη, ιδίω όσον αφορά ε, τη χειρολογική απαιτήση του δευτέρου κεφαλαίου, καθώ επίση και ε, το Capital Guidance Οπότε θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να υπάρχει ομοιογένεια σε πρακτικές και πρότυπα. Επίσης έχουμε υποβάλει συγκεκριμένα σχόλια για κάποια ζητήματα τα οποία πέρασαν από τη διαβούλευση. Περαιτέρω διαβήματα θα πρέπει να γίνουν ούτω ώστε να έχουμε μεταρρύθμιση στην εποπτεία, στην χρηματοοικονομική δραστηριότητα για να δούμε τι θα γίνει πέραν από τους κινδύνους για όλους τους συλλαβισμούς κινδύνους και να κάνουμε κάποια ανάλυση ε, των κεφαλικών στοιχείων τρίτου επίπεδου. Ε, λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει bail-in ε, το οποίο να υλοποιείται, ολοκληρώνεται. Θα πρέπει επίσης να κάτσουμε και να δούμε προσεκτικά τι επιλογές υπάρχουν και τι γίνεται όσον αφορά την κοινωτική νομοθεσία και να δούμε τι εργαλεία υπάρχουν, ιδίως όσον αφορά την εκαθάριση τραπεζών και θα πρέπει πάντοτε να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας της δικαιοσύνης και της ευελιξίας, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο και ποτέ να μην ξεχνούμε ότι θα πρέπει να προστατεύουμε την χρηματοοικονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα. Τέλος, στην έκθεση τονίζουμε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η τραπεζική ένωση. Και το Κοινοβούλιο επίση χαιρετίζει την τελευταία νομοθετική δέσμη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτέ τι προτάσει που υπευλήθησαν και το ότι δεσμεύτηκε η Επιτροπή να συγκρατήσει τον ε, συστημικό κίνδυνο. Επίση, ε, λέμε ότι θα πρέπει να προχωρήσει η νομοθεσία και γι' αυτό και τονίζουμε ότι η συρρήγνωση του κινδύνου είναι μια ευρύτατη έννοια, η οποία αναφέρεται σε διαφορετικά πολλά μέτρα. Και όσον αφορά την έκθεση στον κίνδυνο και σχετικά με τις αποφάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας ότι δηλαδή κάθε αλλαγή θα πρέπει να αξιολογείται και ότι μέσω πρόθεσμα πρέπει να γίνεται αναθεώρηση στα πλαίσια των διεθνών φορέων της εποπτείας της Επιτροπής της Βασιλείας και δεν θα πρέπει να φυγεί η σταθερότητα και η οικονομία των κρατών μελών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γκουαλτήρη λέει ο Πρόεδρος και τώρα τον λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ κύριε Χίλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και τον Ρομπέρτο Κουαλτιέρη για αυτό το ψήφισμα για την ε, Τραπεζική Ένωση. Νομίζω ότι ε, με, εξαιρετικό τρόπο μας υπενθύμισε όλα τα επιτεύγματά μας ε, κατά τη διάρκεια των εργασιών μας για να ξεπεράσουμε τα, το, τα τελευταία χρόνια το, το ελληπές κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτήν είναι αρχιτεκτονική, είναι απαραίτητη η Τραπεζική Ένωση, είναι ο νέος επιπτικός μηχανισμός, νέος μηχανισμός ε, ήδη έχουν καθιερωθεί και εύκολα μπορεί κανείς να ξεχάσει ότι η μετάδοση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό έγινε μόλις πριν από ένα χρόνο ή για το Συμβούλιο Εξυγίανσης ε, ε, λειτουργικό ήταν μόνο από τον Ιανουάριο του 2016. Τεράστια άλματα έχουμε κάνει σε χρόνο ρεκόρ και έτσι έχουμε ενισχύσει ε, την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθιστώντα ισχυρότερε και προστατεύοντα έτσι του φορολογούμενου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη τη Επιτροπή, τα μέλη του Κοινοβουλίου και του προκατόχου μου για το ρόλο του ε, σε αυτό το τομέα. Ε, καλύπτονται πάρα πολλά και διαφορετικά ζητήματα μέσα στην έκθεση. Επιτρέψτε μου να ασχοληθώ μόνο με τα βασικά ζητήματα που σχολίασε ο κύριο Γκουαλτιέρη. Συμφωνούμε ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και φυσικά στο ιστορικό των κρατών μελών θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που εξακολουθούν να βαραίνουν τμήματα του τραπεζικού τομέα. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι αναλογική η νομοθετική ρύθμιση που θα αποφασίσουμε ότι θα λαμβάνει υπόψη τα διάφορα επιχειρησιακά και τραπεζικά μοντέλα και φυσικά θα τηρούνται οι κεφαλιακές απαιτήσει κυρίως για τα μικρά πιστοτικά ιδρύματα. Και αυτό θα δούμε όταν αναθεωρήσουμε την οδηγία CRR για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Ε, θα πρέπει όμως ε, να βάλουμε τα δυνατά μας ε, ούτως ώστε να υποστηρίξουμε ταυτόχρονα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε προγράμματα υποδομής. Πέρα από την ενίσχυση της Τραπεζικής Ένωσης βλέπουμε μέσα στην έκθεση και στη δική μας πρόταση βασική εστίαση είναι να δημιουργήσουμε μέχρι το 2024 το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων ΕΝΤΙΣ ως τμήμα του συνολικότερου προγράμματος ενίσχυσης της Τραπεζικής Ένωσης. Έτσι θα έχουμε το τρίτο πυλώνα, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί με την δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης. Έτσι θα έχουμε μια ισόρροπη προσέγγιση, χάρη στην οποία θα περιορίσουμε τους κινδύνους και θα αμοιβεοποιήσουμε τους κινδύνους. Είναι ζωτική σημασία να προωθήσουμε εκ παραλληλού τα δύο τμήματα αυτή τη πολύπλοκη εξίσωση. να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση ούτω ώστε η οδηγία για την, την εξηγία των τραπεζών και για τι κεφαλικές απαιτήσει να μεταφερθούν πλήρω στην εθνική νομοθεσία. Σχεδόν τα έχουμε καταφέρει γι' αυτό αυτό και στη συνέχεια ε, θα δούμε ποιες είναι οι βασικές διαφορές στην αφαιρεγγιότητα και στα συστήματα προορή εξυγίανσης ε, και πρώτο τέλος του 2016 θα κάνουμε μια πρόταση ούτω ώστε να έχουμε το πρότυπο TILAC ε, με τρόπο που να λειτουργεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από λίγο τόνισε ο κύριος Γκουαλτιέρη τις ανησυχίες που έχει για τις κεφαλιακές απαιτήσει των τραπεζών για τον πυλώνα 2 και τη σχέση που υπάρχει με τα αποθεματικά έκτακτη ανάγκης ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορές ως προς την εφαρμογή των κανόνων από τις εποπτικές αρχές ε, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο μου έχουμε δρομολογήσει τη διαδικασία εξέτασης από κοινού με τα κράτη-μέλη και με θεσμικά όργανα όπως το Κοινοβούλιο και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, ούτως ώστε η νομοθεσία να λειτουργήσει όπως αρχικά είχε προβλεφθεί. Θα πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στους κανόνες ε, του πυλώνα 1 που ισχύει για όλες τις τράπεζες και τις απαιτήσεις του πυλώνα 2 που ναι, είναι για συγκεκριμένα πιστοτικά ιδρύματα και είναι συνάρτηση του επιπροσθέτου κινδύνου που ενδεχομένως έχουν τα χαρτοφυλάκια κάποιων μικρότερων πιστοτικών ιδρυμάτων. Ε, ε, εκτιμώ όλα αυτά που είπατε και φυσικά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για αυτό τόσο σημαντικό ζήτημα. Αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα που τράβηξαν την προσοχή μου στην έκθεση του κ. Γκουαλτιέρη. Είναι γερά τα θεμέλια από τον οποίο θα οικοδομήσουμε τη μέλος αρχιτεκτονική και είμαι αισιόδοξο ε, σε σχέση με τις ευκαιρίε που έχουμε να χτενίσουμε περιττέρω την νομοθεσία, ούτω ώστε να υλοποιήσουμε του στόχου μα για τη μακροληπτική εποπτεία. Ταυτόχρονα όμω να τονώσουμε και την ανάπτυξη, να προστατεύσουμε τι επενδύσει Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε, Επίτροπε Χίλε. Τώρα θα ακούσουμε του εκπροσώπου των πολιτικών ομάδων και μετά θα αρχίσει και η διαδικασία ε, των γαλάζιων καρτών στα πλαίσια της συζήτηση από πλευράς ε, του ΕΛΚ η κυρία Πάνοβα. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα σημαίνει ανάπτυξη, δουλειέ και σταθερότητα. Πρόσφατα είδαμε τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε κάποια κράτη-μέλη να γνωρίζουν ε, ε, χρηματοπιστωτικές αναταράξεις. Αυτό δείχνει ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Η έκθεση ε, έχει τη σωστή κατεύθυνση και το σωστό τόνο για τις μεταρρυθμίσεις στο τραπεζικό σύστημα. Και είναι σημαντικό ότι ζητεί να μειωθεί ο ηθικός κίνδυνος. Το κόστος για τις αφαιρεγγιότητες ε, και τη χρεοκοπία των τραπεζών θα πρέπει να αμοιβιοποιηθεί αλλά ε, να συγκρατηθεί ταυτόχρονα. Ε, δεν ε, χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα, γι' αυτό ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει τέτοια μέτρα και τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τους κείμενους κανόνες. Η ε, του τραπεζικού τομέα θα πρέπει να συνοδεύεται από νομική ασφάλεια. Αυτό ζητούμε να διευκρινιστεί η νομοθεσία MTA για να μπορούν οι τράπεζες να σέβονται ε, τις κεφαλαϊκές απαιτήσει και του πρώτου και του δευτέρου επίπεδου. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μειωθεί το δημόσιο χρέο και να υπάρχει μια ε, ισόρροπη προσέγγιση προς τον τρίτο ε, πυλώνα. Γι' αυτό ζητούμε ένα σύστημα με προληπτική υποπτία είναι συντριπτική η πλειοψηφία στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, ελπίζω και στην Ολομέλεια, για να αρχίσει ένα σημαντικό διάλογο που θα μα βοηθήσει να οικοδομήσουμε ε, όσο γίνεται καλύτερα μια τραπεζική ένωση. Ευχαριστώ από σοσιαλιστέ και δημοκράτε, η κυρία Φεραίρα, για 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το, η μόνη ολοκλήρωση που έχουμε καταφέρει από το 2008 στην Ευρωζώνη. Έχουμε την έκθεση των τεσσάρων Προέδρων και της ε, Επιτρόπου Τάισεν και καταλήγει στο ότι η Τραπεζική Ένωση Επαναλαμβάνω, όπω λέει η έκθεση του 2015 είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για το χρηματοπιστωτικό ευρωπαϊκό σύστημα. Και αυτό προέκυψε ε, σαφώς κατόπιν των με το Κοινοβούλιο που είναι ε, πρωτοπόρο. Και έχουμε επομένως αυτό το σύστημα εποπτείας το οποίο ε, ολοκληρώθηκε πάρα πολύ νωρίς. Πρόκειται επομένως για μια υπόθεση υψηλού κινδύνου. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις λεπτομέρειες αυτού του συστήματος θα πρέπει να υπάρξει αμοιβή εμπιστοσύνη. Υπάρχουν παρόμοια συστήματα και στη Γερμανία αλλά και στις ΗΠΑ. Είναι θέμα ασφάλιση των καταθέσεων. Αυτό είναι προϋπόθεση για να υπάρχει η οικονομική σταθερότητα. Εάν δεν μπορέσουμε όλα αυτά τα στοιχεία να τα υλοποιήσουμε και κυρίως στον τρίτο πυλώνα, ιδίως το θέμα της ασφάλισης των καταθέσεων με το έντις, αλλά να μπορέσουμε επίσης να αναθεωρήσουμε το SMUS θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους κινδύνους του να διαλυθεί το σύστημα, καταρρεύσει. Γιατί μπορούν να γίνουν παράγοντε ανισορροπία και όχι σταθεροποίηση πλέον, αν δεν ολοκληρωθεί η προσπάθεια μα. ξέρετε ότι όταν ένα γλυκό το έχουμε ψήσει μέχρι τέλου, είναι μια ευχαρίστηση. Αν το έχουμε μίσο ψήσει, τότε θα μα πέσει βαρύ στο στομάχι. Ε, Φωνστόρ και 1,5 λεπτό από του συντηρητικού. Herr Κύριε Πρόεδρε, σήμερα μιλούμε για την Τραπεζική Ένωση που μέχρι τώρα έχει δύο στοιχεία. Η αμοιβιοποίηση του κόστους για την εκαθάριση ε, ε, τραπεζών που χρεοκοπούν και την πληρώνουν πάλι φορολογούμενοι, ιδιαίτερα οι Γερμανοί. Και το δεύτερο είναι μια ενιαία τραπεζική εποπτεία που δεν λειτουργεί. Και ακόμα χειρότερο, η τραπεζική εποπτεία και η νομισματική πολιτική τώρα αναμειγνύονται. Δεν έχουμε ανεξάρτητη πολιτική πλέον νομισματική. Το έχει επικρίνει ο κύριο Σόιμπλε, χριστιανοδημοκράτη, και η αλλαγή ζήτησε τροποποίηση των συνθήκων. Αγαπητοί συνάδελφοι της Τσέντεου, έχω κάνει τροπολογία στην Επιτροπή για να διαχωριστεί η εποπτεία από την νομισματική πολιτική και εσείς δυστυχώς δεν το υποστηρίξατε. Και τώρα έρχεται ένα τρίτο στοιχείο που είναι λέει η κοινή ασφάλιση και προστασία των καταθέσεων. Αγαπητοί συνάδελφοι Τσέντεου, Τσέσου, S5, FTP από τη Γερμανία. Σήμερα τι συζητούμε οι Γερμανοί καταθέτες και αποταμιευτέ θα πρέπει να πληρώνουν τα σπασμένα για ξένες τράπεζες ε, Τέρματα τα κηρύγματα και τα ωραία λόγια σήμερα θα πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας και εγώ ζήτησα ονομαστική ψηφοφορία για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια Προστασίας Καταθέσεων για να καταλάβουν οι ε, εκλογής στα τρία κρατήδια που έχουν εκλογές στη Γερμανία την Κυριακή ε, ποιος ε, λέει τι για να πάει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Το κόμμα μου ο ΑΕΦΤ είναι κατά της πρότασης αυτής. Η κυρία Γκουλάρ για δύο λεπτά από τους φιλελευθέρους. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Επίτροπε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω την Ένωση για την Τραπεζική, τη ψήφισμα για την Τραπεζική Ένωση και να πω ότι δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε για κομματικού σκοπού και για την προεκλογική μα εκστρατεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα και ε, επιτέλου μπορούμε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα. Ευχαριστούμε, Ρομπέρτο, για τη δουλειά που έκανε. Ε, μια σφαιρική εικόνα για τα όσα έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Κατά πάσα πιθανότητα, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια και μοναδική επιτυχία, πραγματική επιτυχία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μεγάλο άλμα για τα ουσιαστικά ουσιαστικά και σημαντικά προβλήματα. Δεν θέλω να επανέλθω αυτά που ήδη ακούσαμε. Θέλω και εγώ να ασχοληθώ με το σύστημα ΕΝΤΙΣ, γιατί είμαι και σκιώδη για το σύστημα, δηλαδή Ευρωπαϊκό Σύστημα κατάσταση εγγύσεων, ε, ε, ε, των καταθέσεων, συγγνώμη. Ε, χρειαζόμαστε αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτό το κείμενο πραγματεύεται πολύ σημαντικά ζητήματα, διότι εγώ αρνούμαι να ε, επανεθνικοποιούμε ε, τέτοια ζητήματα. Δηλαδή σε όλες τις χώρες είναι σημαντικό να ε, κατοχυρώνουμε, να εγγυόμαστε τις καταθέσεις. Το εξίσου σημαντικό είναι και το ζήτημα της υγείας του τραπεζικού τομέα μέσα στην Ευρωζώνη. Είναι τόσο στενή η δεσμή που μας ενώνουν που πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Δεν θα πρέπει αντιμέτωποι με ένα να θεωρούμε ότι μπορούμε εν μία νυχτή να τροποποιήσουμε την κατάσταση. Η εμπιστοσύνη λοιπόν μεταξύ μας και τι μπορούμε να κάνουμε. Επίτροπε, από τις πρώτες ε, συζητήσεις που κάναμε για αυτό το θέμα, έκρινα ότι είναι σημαντικό να ε, ε, παίξει το ρόλο του θεματοφύλακα των συνθήκων ε, πλήρωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα διότι το σημαντικό είναι να γίνει καλή δουλειά και αυτό μπορεί να χρειαστεί χρόνο για να σημειώσουμε και πάλι επιτυχία. Ξαναλέω πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και σας ευχαριστούμε για αυτή την πρόταση γιατί πρόκειται για την, ε, ε, το τρίτο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης. Ευχαριστούμε Κάρια. Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα κυρία Κάρη, έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν διασώσαμε τις τράπεζες κατά την ε, χρηματοοικονομική κρίση, αυτό έγινε με λεφτά των φορολογουμένων. Γι' αυτό γιατί θυμάστε ήταν πολύ μεγάλες για να χρεοκοπήσουν αυτές οι τράπεζες και θα είχαν παρασύρει και την υπόλοιπη κοινωνία στη χρεοκοπία. Επομένως ένα από τα πρώτα μας βήματα είναι να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους φορολογουμένους για την επόμενη χρήση. Να κάνουμε δηλαδή τόσο μεγάλες τις τράπεζες που να μην, υπάρχει πρόβλημα. Όμως δεν κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρασαν 8 χρόνια από την αρχή της ε, κρίσης και ο τραπεζικός τομέας έχει μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και γίνει ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει νομοθεσία που να λαμβάνει υπόψη αυτές τις τράπεζες τις πολύ μεγάλες για να χρεοκοπήσουν και ακόμα μπορούν να γίνουν μεγαλύτερες. Οπότε ε, έτσι ε, δεν θα υπάρχει άλλη τραπεζική κρίση. Να, έχουμε τραφεί την πρώτη έκθεση, την ετήσια για τις τράπεζες. Θα πρέπει επομένω στο θεματολόγιο να μπει και αυτό το θέμα των μεγάλων τραπεζών, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το έχει λάβει αυτό υπόψη και ο Μάριο Ντράγκη και αυτός ανήκει σε αυτή την ομάδα, στην ομάδα αυτών των 30 ε, μεγάλων τραπεζών. Μα είναι μέλος επομένως μιας λέσχης διοικητών τραπεζών, προέδρων τραπεζών, μα αυτούς έπρεπε να τους εποπτεύει. Δεν νομίζω ότι του εποπτεύει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η έκθεση ότι είναι αξιόλογη και επικριτική. Δεν την ψηφίζουμε. Για του πρασίνου τώρα έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Γκίγκολτ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, καταρχά θέλω να πω ότι είναι αρκετά θλιβερό να βλέπουμε ότι γίνεται μια απόπειρα με ανακρίβειες να κάνετε κομματική πολιτική και προεκλογική. Ακριβώς το θέμα δεν είναι οι φορολογούμενοι να ε, έχουν την ευθύνη για την προστασία των καταθέσεων ούτε για την εκαθάριση των τραπεζών, αλλά η Τραπεζική Ένωση εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το σκοπό να προστατεύει τους φορολογουμένους, γιατί στο μέλλον οι πιστωτές θα έχουν την ευθύνη και εφαρμόζεται η αρχή τη ελεύθερη αγορά. Είναι ανακρίβειε αυτά που λέτε κύριε Φωνστόρχ και κινδυνολογείτε και δυστυχώ και στη Γερμανία πρέπει να σα ανεχόμαστε. Ε, Εκπλήσωμαι ε, που εκφράζεται τέτοια κριτική από την αριστερά για την έκθεση. Θα χαιρόμουν αν ήσασταν παρόντες στις διαπραγματεύσεις και λέγατε τη δική σας θέση εκεί στους κοιόδης ηγητές. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε, να έρχεστε στην Ολομέλεια εκ των υστέρων για να κάνετε κριτική, ενώ στις διαπραγματεύσεις που έγιναν συλλογικά υπό την ηγεσία του κυρίου Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη απουσιάζατε. Και αυτά θα πρέπει να τα λέμε. Και να πω το εξή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλωσορίζω και χαιρετίζω πολλά από τα όσα εφαρμόζετε Θα παρακαλούσα το εξή. Στην έκθεση υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που δεν έχουν μπει ακόμα στο πρόγραμμα εργασία σα. Λίγα είπατε σχετικά, κύριε Χιλ. Τι κάνετε κατά τον. Ε, σχεδόν τραπεζών. Ε, το παράλληλο σύστημα, τι γίνεται, το, με το αρμπιτράζ ε, και την διαιτησία και τη, σε ασφαλιστικές εταιρείες σε σχέση με τις τράπεζες και με απασχολεί πάρα πολύ το εξής. Υπάρχουν διάφορα μηνύματα που λένε να μειωθεί το ίδιο κεφάλαιο ως ποσοστό. Θα το σταματήσετε αυτό γιατί δεν επιτρέπεται να επαναλάβουμε σφάλματα του παρελθόντας Ευχαριστώ. Διαδικαστικό έχετε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, ο Διερμηνέας κατά την ομιλία της κυρίας Γκίγκολτ είπε ότι η κυρία Φανστόρκ είπε κάτι το οποίο είναι αναλυθές στα αγγλικά. Αυτό σημαίνει ότι είπε ψέματα. Η κοινοβουλευτική αγωγή επιτρέπει το να αποκαλεί κάποιον συνάδελφο, κάποιος ψεύτη. Μήπως έκανε λάθος ο ή η η Δεν το είπε αυτό η κυρία Γκίγκολτ. Οπότε τι θα κάνω. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, θα το κοιτάξουμε. Ε, βάλει. 1,5 λεπτό για το EFTD. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να πω στην κυρία Γκίγκολ το εξή ότι οι Γερμανοί φορολογούμενοι είναι ακόμα πιο εκτεθειμένοι παρά τους δύο πρώτους πυλώντες γιατί όταν έγινε ο πρώτος πυλώνας κύριε Χιλ τότε είχαμε μια διάκριση, έναν διαχωρισμό. Είχαμε παγκόσμιες τράπεζες που μπορούσαν να κερδοσκοπήσουν, να σπεκουλάρουν και κατόπιν ε, κάνατε αυτή την... Ε, Μα δεν είναι κανονιστής διαχωρισμός. Ε, για ακούστε τι, τι λέει ο κόσμος και κατόπιν φτιάξατε τον δεύτερο πυλώνα με την έννοια του τρέχοντος λογαριασμού ως επένδυσης και λέτε ότι τώρα θα έχετε το όριο των 100.000 αυτό δεν λέει τίποτα. Και επομένως αυτά τα 100.000 ευρώ και ότι υπάρχει παραπάνω πάνε. Οπότε ε, έτσι θα πρέπει να δούμε ποιος είναι τελικά αυτός που τελικά θα διασώσει την κατάσταση, τη τελευταία καταφυγή όπως λένε, θα πρέπει να σκεφτείτε ποιες είναι όχι οι αιτίε, αλλά οι συνέπειες της κρίσης. Αυτό είναι ένα παράδοξο. Είναι, είναι κάτι το τερατώδες αυτή η αστάθεια του ζήματος είχαμε 40% μείωση των αποθεμάτων την πρώτη πρώτο. Γι' αυτό και δεν λειτουργεί το σύστημα. Συνέχεια συζητάμε για ε, τις πιστώσει, συζητάμε για την ασφάλιση των καταθέσεων και δεν μιλάμε για τα τραπεζικά προϊόντα. Είδατε τι έγινε με τα derivatives στην Γαλλία. Θα έπρεπε στον πρώτο πυλώνα να κάνετε αυτόν τον διαχωρισμό των τραπεζών. Ευχαριστούμε κύριε Βάλλη και τώρα για την ENF έχει το λόγο ο κύριο Μόνο. Επίτροπε Πρόεδρε, αν έντερ να κάνω τον απολογισμό τη Τραπεζική Ένωση για το 2015, θα έλεγα ότι η θεσμική σα απάτη για να ξανασώσετε και πάλι το τραπεζικό λόμπι λειτουργήσε καταπληκτικά για εσά μέχρι στιγμή. Η νομοθεσία, τη νομοθεσία τη εικόνα στι πλάτε του οι φορολογούμενοι, γιατί έγινε τον Αύγουστο με διάταγμα η έγκριση τη Τραπεζική Ένωση, την ώρα που οι Γάλλοι ήταν στην παραλία. Όταν λοιπόν θα έχουμε αφαιρεγκιότητα, θα καταρρεύσει το σύστημα, στην παγίδα θα πέσουν οι φορολογούμενοι και θα πληρώσουν με τις αποταμιεύσεις τους ε, την επαναχρηματοδότηση της ε, τράπεζας. Ε, αυτό το σύστημα της ΕΚΤΕ, αυτός ο απολυταρχισμός, ο χρηματοπιστωτικός απολυταρχισμός για να σωθεί και πάλι το ευρώ είναι που καταγγέλουμε. Ο τρίτος πυλώνος προβλέπεται 8 χρόνια, δεν είναι δημοκρατικός και δεν πρόκειται ποτέ να θεσπιστεί γιατί δεν το θέλει η Γερμανία. Είδαμε με την πτώχευση πριν από λίγα χρόνια των τεσσάρων περιφερειακών τραπεζών της Ιταλίας ότι δεν εφαρμόζεται ε, ο κανονισμός, ε, ε, καταστρέφονται οικονομικά και ορισμένοι αυτοκτονούν κιόλα από τους πελάτες της τράπεζας. Είναι ο κίνδυνος, απειλεί τη δημοκρατία και η μόνη λύση είναι να, να έχουμε την... την... να σταματήσουμε με αυτές, με αυτές τις ουτοπίες της Καθολικής Τράπεζας για το μόνο που κάνουμε είναι να διωγγώνουμε τους κινδύνους και τα προβλήματα. Οι κυρίαρχοι λαοί της Ευρώπης θα στραφούν γύλη κατά την, ε, το δικό σας οικοδόμημα που απειλεί τη δημοκρατία. Ευχαριστούμε. Ε, από τους μη γραμμούς ο κ. Ζεργιανόπουλος, ένα λεπτό παρακαλώ. Ισχυρίζεστε ότι η Τραπεζική Ένωση εξηγαίνει τις τράπεζες χωρίς να επιβαρυνθούν τα λαϊκά στρώματα, αλλά δίθεν μέτοχοι και μεγαλοκαταθέτες. Είναι ψέματα. Για παράδειγμα, τα κόκκινα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κρίσιμη πτυχή τη Τραπεζική Ένωση, αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα των τριών μνημονίων, αποτέλεσμα τη ανεργία και τη γενικευμένη λαϊκή φτώχεια η αξιολόγηση κουαρτέτου και κυβέρνηση σύριζα τα οδηγεί σε διεθνή κερδοσκοπικά φαντ σφίγγοντας περισσότερο τη θηλιά και εντείνοντας το κυνηγητό στα λαϊκά νοικοκυριά. αυτά πλήρωσαν με μνημόνια την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών τώρα θα πληρώσουν και την εξυγίασή του με την απώλεια τη στέγη του με χιλιάδε πληστηριασμού που απελευθερώθηκαν. η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν έρχεται όπω θέλετε. οι Τράπεζέ σα έχουν πρόβλημα γι' αυτό συγκεντρώνεται ενισχύεται το τραπεζικό σύστημα η εναλλακτική χρηματοδότηση από την ένωση κεφαλαίου ή από τι ενισχυόμενε ιδιωτικέ ασφαλιστικέ που σαν τα κοράκια εκμεταλλεύονται την καταδάφιση τη κοινωνική ασφάλιση. δηλαδή και την κρίση και την ανάκαμψη του καπιταλισμού θα πληρώσει ο λαό αν δεν επιλέξει το δικό του δρόμο για την εξυπηρέτηση των δικών του σύγχρονων αναγκών ενάντια στο κεφάλαιο και την εξουσία του. Ευχαριστώ κύριος Μπάλτς για λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, η έκθεση για την Τραπεζική Ένωση ρίχνει μια ματιά στο περασμένο έτος και στους τρεις πυλώνες ε, της Τραπεζικής Ένωσης χρειάζεται δουλειά για να ολοκληρωθεί το έργο. Πριν όμως οικοδομήσουμε την ε, Τραπεζική Ένωση και χτίσουμε περισσότερο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η οικοδόμηση τη προηγούμενη φάσης και τα κράτη-μέλη καλούνται να υλοποιήσουν ε, τις υποχρεώσεις τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει την απαραίτητη πίεση. Διότι Εάν δεν είναι σταθερά τα θεμέλια της Τραπεζικής Ένωσης, ό,τι και να οικοδομήσουμε πάνω θα ε, είναι σε σαφρά θεμέλια. Βλέπω ε, όλο και, με όλο και περισσότερη ανησυχία να γίνεται λόγος για μεγαλύτερη ευελιξία και αμοιβαιοποίηση. Κυρίες και κύριοι, ας εφαρμόσουμε πρώτα τα όσα ε, αποφασίσαμε, ε, γιατί ε, αυτά για τους πιστωτές δεν είναι κάτι που θα πρέπει να βαρύνει τους πολίτες. Χρειάζεται με ευθύνη ε, και συνέπεια να προστατεύουμε τους φορολογουμένους, να έχουμε ένα σύστημα συμμετοχής των ε, πιστωτών και ένα bail-in. Ε, θα πρέπει τώρα να υλοποιήσουμε όλα αυτά που αποφασίσαμε για περαιτέρω μείωση του ηθικού κινδύνου που είναι απολύτως απαραίτητη. Γι' αυτό κύριε Επίτροπε ζητούμε και νομοθετικές προτάσεις για να υπάρχει μια σταθερή τραπεζική ένωση αποτελεσματική για την οποία θα συνεργαστούμε αλλά για να γίνει αυτό απομένει ακόμα πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Μπάλτς, ο κύριος Βάλλη έχει μπλε κάρτα, τη δέχεστε. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπάλτς για την απάντηση. Ενημερωτικά ο κάθε αγορητής δέχεται μία επερώτηση. Θα γίνουν οι ψηφοφορίε το απόγευμα. Κύριε Βαλή, για το λόγο. Ευχαριστώ για την απάντηση που θα μου δώσετε, κύριε Μπάλτ. Είπαμε ότι έχουν θεσπιστεί αυτοί οι κανόνε. Και το 2013 είπαμε ότι δεν μπορούσαν πια να υπάρχουν κρατικέ επιδοτήσει. Και τελικά είχαμε τέσσερι τραπέζε στην Ιταλία τώρα, ε, επί των οποίων πάρα πολύ αυστηρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε για πετε μα, γιατί δεν υπήρχε η ίδια αυστηρότητα και όσον αφορά τι έγινε και σε εκείνη, για εκείνη την γερμανική τράπεζα ήταν αυστηρή με εμά η Κομισιόν και όχι με τη Γερμανική Τράπεζα. Σε εκείνη δώσανε τρία δις ε, επιδότηση. Γιατί άλλοι κανόνες ισχύουν για τη Μεσόγειο. Κάνει ό,τι θέλει η Γερμανία. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό. Καταρχάς δεν κατάλαβα πάρα πολύ καλά από τη διερμηνία τη ρωτήσατε. Θέλω να πω ξεκάθαρα ότι θεωρώ απολύτως σωστή την αυστηρή ε, μεταχείριση των Ιταλικών τραπεζών και η ίδια στάση θα πρέπει να ισχύει και για άλλους. Αγαπητέ συνάδελφε Βάλλη, για αυτό το θέμα απευθυνθείτε στον Επίτροπο τον κύριο Χιλ, ο οποίο είναι και παρόν άλλωστε και μπορεί να μιλήσει εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ πιστεύω ότι είχε απολύτω δίκιο στάση τη απέναντι στι Ιταλικέ ε, τράπεζε η Κομισιόν. Ο κύριος Φον Βάιτσεκερ για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Ρομπέρτο Κουαλτιέρη για την ε, εξαιρετική του έκθεση. Βασικό μήνυμα ποιο είναι. Ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση και όχι μισό μισοάδιο διότι έχουν επιτευχθεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά μόνο μισό γεμάτο λέγω, διότι απομένουν ακόμα περισσότερα για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα. Και ακριβώς επειδή είναι μισογεμάτο το ποτήρι, αυτό που ε, προτείνει ως αναθεώρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ρυθμιστικά δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως οπισθοδρόμηση, αλλά μια αναθεώρηση για να γεμίσουμε το υπόλοιπο που απολύπτεται. Ε, στην Τραπεζική Ένωση υπάρχει πρόβλημα ε, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί. Η κεφαλαιοποίηση παραμένει άνηση και ιδιαίτερα για τις συστημικές τράπεζες δεν είναι απολύτως ικανοποιητική πάντοτε. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους ε, για τις πρόσφατες αναταράξεις στην αγορά. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διαρθρωτική μεταρρύθμιση των τραπεζών θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά και να μην αποδυναμώνεται. Θα πρέπει ε, το 8% του μπέιλιν να μην ε, εμποδίζει, ε, αλλά να προστατεύει ουσιαστικά τους φορολογουμένους. Ε, θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα προστασίας των καταθέσεων ε, ευρωπαϊκό, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και γνωρίζοντας ότι αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από τη μείωση του ηθικού κινδύνου. Σημαντικό είναι να μην εκτίθενται οι τράπεζες υπερβολικά στο δημόσιο χρέος. Είναι λοιπόν καλή έκθεση ε, του Γουαλτιέρη για να δούμε πώς θα γεμίσουμε ένα μισογεμάτο ποτήρι. Έχετε μπλε κάρτα. Από τον κύριο ε, Γουλφ. Τη δέχεστε. Thank Ευχαριστώ. Κύριε Βάιθτσα, κύριε. Απλή ερώτηση. Έχουμε αυτή την έκθεση για την Τραπεζική Ένωση και εσεί. τι πιστεύετε, υπάρχει μία μόνο μέθοδος εποπτείας των τραπεζών στην Ένωση ή θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλες μεθόδους και εναλλακτικέ για να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό, το πρόβλημα στην απασχόληση εκτός από την Τραπεζική Ένωση. Η βελτίωση της Τραπεζικής Ένωσης δεν είναι ε, ούτε ικανή ούτε η αναγκαία μοναδική συνθήκη για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το ώστε να έχουμε μακρόπνοη εύρυθμη λειτουργία των οικονομιών μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Και όπως γνωρίζετε, δεν ανήκουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής στην Τραπεζική Ένωση. Ούτε όλα τα μέλη της ε, Ευρωζώνης. Ε, γι' αυτό και λέμε ότι υπάρχει μια πρόκληση σε σχέση με τα σημερινά προαπαιτούμενα ως προς την τραπεζική νομοθεσία και σε σχέση με το κοινωνικό δίκαιο της ενίας αγοράς. Γι' αυτό ε, και παρουσιάζει τόσο ενδιαφέρον η δουλειά της Επιτροπής μας. Λοιπόν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή για την Τραπεζική Ένωση περιλαμβάνει κάποια πολύ καλά στοιχεία. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι είναι πολύ επικριτική ματιά για τις ε, ε, δοκιμασίες αντοχής, τα stress τεστ για τις μεγάλες τράπεζες. Ακόμα και η δέξια η τράπεζα αυτή ε, έχει περάσει το τεστ στο παρελθόν και όλοι ξέρουμε τι έκβαση είχε. Αν θέλουμε οι τράπεζε στην Ευρώπη να είναι αποτελεσματικέ, χρειάζεται περισσότερο έλεγχο, ισχυρότερο και συχνότερο. Στο μέλλον θα πρέπει να το προσέξουμε στο Κοινοβούλιο και να το συζητήσουμε ας πούμε το θέμα της εγγύησης των καταθέσεων που μας απασχολεί σήμερα είναι πάρα πολύ σχετικό. Τέλος, πρέπει να πω ότι λυπάμαι για το εξής. Σε κάποια ε, θέματα η έκθεση τα λέει πάρα πολύ ρόδινα. Για παράδειγμα, τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Που οι τράπεζες έχουν τρομερή έκθεση, ιδιαίτερα στην Νότια Ευρώπη. Θα πρέπει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 και δείχνουν λαϊκισμό, δημαγωγία ή άγνοια σε σχέση επίσης και με το τι θα πει η δημοκρατία γιατί αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι η Τραπεζική Ένωση ίσως είναι ό,τι πιο σημαντικό και ουσιαστικό έχει γίνει σε σχέση με την λαϊκιστική επανεθνικοποίηση των όσων αφορούν τους Ευρωπαίους και έγινε τα τελευταία χρόνια για να εξασφαλίσει την ευημερία στις μέλουσες γενιές Ευρωπαίων. Ξέρω ότι προχωράει, ξέρω ότι είναι κάτι τεχνοκρατικά προχωρημένο, εδώ όμως μιλούμε για πολιτική και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ότι προχωράμε προς περισσότερη ασφάλεια και δημοκρατικότητα και αυτό γίνεται με fair play, γίνεται με ταχύ αλλά παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει μεγάλη προσοχή γιατί αλλιώς θα αρχίσουν οι σιρήνες της επανεθνικοποίησης. Κύριε Καλβέντη, υπάρχει μια υπερώτηση από τον κύριο Τσάνι. Δέχεστε. Κύριε Τσάνι, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, συμφωνώ όταν λέτε ότι πρόκειται για μένα μεγάλο επίτευγμα, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Θα ήθελα να ξέρω εάν θεωρείται ότι ε, πρόκειται για μεγάλη επιτυχία ε, όταν δεν έχουμε εγγύηση των καταθέσεων. Δεν υπάρχει, δίκτυα δίκτυο ε, ασφαλείας. Excuse, Presidente. Penso... λέει ο κύριο Καλβέτ. Νομίζω ότι είναι κάτι το πετυχημένο στην έμπνευσή του αλλά τώρα είμαστε στην αρχή της διαδρομής, άρα θα πρέπει να προχωρήσουμε καλύτερα και πιο γρήγορα. Κύριε Ούρμπαν Κρέσπο, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε συναδελφοί, 8 χρόνια από τότε που άρχισε η κρίση, 700 δις έχουν πάρει οι τράπεζες από το δημόσιο. Δηλαδή σαν να έχουν πάρει πέντε ενωσιακούς προϋπολογισμούς. Πέραν αυτό όμως οι μεγάλες τράπεζες του Βορρά σήμερα είναι η μεγάλη μαύρη τρύπα στην Ευρώπη. Και μιλάμε για 60 εκατομμύρια. Πέντε φορές το γερμανικό ΑΕΠ. Και οπότε τα ευρωπαϊκά δεσμικά όργανα είναι άχρηστα. Δεν μπόρεσαν τις μεγάλες τράπεζες ε, να τις ε, ρεγουλάρουν. Δεν μπόρεσαν να βάλουν σε τάξη τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Όμως ε, τώρα η έλλειψη αξιοπιστίας των τραπεζών αυτών μας οδηγούν σε μια νέα κρίση. Το λέει και η έκθεση ότι ήταν λέει επιτυχία η πρώτη χρονιά της Τραπεζικής Ένωσης. Μα για να ισχύει κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από το να επιβάλλουμε με κάθε μέσον την ε, λιτότητα στις νότιες χώρες και να στέλνουμε το λαό τους στην ε, δυστυχία. Αυτό είναι κάτι σαν ε, ένα πραξικό πείμα όπως έγινε τον Ιούνιο του 2015 στην Ελλάδα το κλείσιμο των, του περιορισμού το, τραπεζικό στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ κακό. Δεν λέει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αγαπητοί μου, αυτά τα θεσμικά όργανα είναι ασκήνιο για την σταθερότητα και την εθνική κυριαρχία στην Ευρώπη. Θα πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση και να αρχίσουμε αυτό να το παλεύουμε τώρα. Δύο λεπτά ο κύριος Γουλφ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, πολλά χρόνια πριν πάμε στο φεγγάρι, πριν από τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο, πριν και από το ε, άρχισε, ε, αναδύθηκε μια νέα αυτοκρατορία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και σκέφτηκαν ότι θέλουμε νέο νόμισμα και νέα τράπεζα, την ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για καλύτερα παραγωγικότητα, μεγαλύτερες θέσεις, περισσότερες θέσεις απασχόλησης, ε, καλύτερες πιθανότητες απασχόλησης για τους νέους. Τι βλέπουμε σήμερα, η ανεργία των νέων σε πολλές χώρες ξεπερνάει το 30%, η παραγωγικότητα μειώνεται, το ΑΕΠ μειώνεται και σήμερα ο κόσμος προχωράει, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ιδέες της όχι το αντίθετο και τεταλαντούχοι άνθρωποι σαν και εσάς, Επίτροπε Χίλε, προσπαθούν να ολοκληρώσουν μια παλιά ιδέα από, τον, ε, από εποχές και να το μεταφέρουν σε ένα σύγχρονο κόσμο. Σκεφτείτε πόσες περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, έχουν ανθούσα οικονομία. Γιατί τα καταφέρουν καλύτερα. Ευχαριστούμε κύριε Γουλφ. Ο ο κύριος ε, Χοκμάρκ ε, θα ήθελε να σας κάνει μια ερώτηση βάσει της ε, μπλε κάρτας. Το δέχεστε πολύ ωραία. Ε, ναι, βλέπω νοσταλγείτε το, την εποχή ε, που έχει παρέλθει και προσοχή γιατί τότε είχε και Vikings. Και όλα τα προβλήματα, αν σας πιστέψουμε, προέρχονται από τις Βρυξέλλες. Για δείτε όμως ποια προβλήματα έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μήπως ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ε, περισσότερα τα προβλήματα ακριβώς για τους λόγους που αναφέρετε. Μήπως ε, δεν χρειαζόμαστε αυτή τη ζούγκλα διαφορετικών νομοθεσιών και χρειαζόμαστε αυτή την ενιαία κάλυψη που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς τι προτιμάτε, μία ζούγκλα ή ένα κοινό κανονισμό ο οποίος τελικά ανοίγει τις αγορές. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο για την ε, απάντηση. Πάντοτε χαίρομαι όταν μου κάνετε ερωτήσεις, ε, κύριο Χέκμα. Το σημαντικό είναι αυτό που λέτε, ζούγκλα. Εγώ μιλάω για ανταγωνιστικέ νομοθεσίε ε, σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ευρωζώνη έχετε υψηλή, έχουμε υψηλή ανεργία, αρνητικό πληθωρισμό, σχεδόν από πληθωρισμό, χαμηλή παραγωγικότητα, όμως χώρε όπω ε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εκτός Ευρωζώνης και έχουν πιο ευέλικτη, πιο ανταγωνιστική βάση και Έχουμε ε, υψηλά αναπτυξιακά επίπεδα, υψηλή παραγωγικότητα, ε, ε, υψηλή απασχόληση σε σχέση με τα κράτη της Ευρωζώνης. Και πρέπει να αναρωτηθείτε το αντίθετο με αυτό το ενιαίο σετ κανόνων. Μήπως έτσι καταστρέφεται την Ευρώπη αντί να έχετε αυτού του ανταγωνιστικού κανόνε που οδηγούν σε εξέλιξη, σε παγκόσμια κλίμακα. Ευχαριστώ. Ρέβεκα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Τραπεζική Ένωση είναι η εκχώρηση ε, εξουσίας στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αν δεν μπορεί κανείς να παίρνει τις αποφάσεις που αφορούν την επικράτειά του και περιμένει μια κεντρική απόφαση από τις Βρυξέλλες. Σα ευχηστώ την προσοχή στο γεγονό ότι η τραπεζική αγορά διαφέρει από χώρα σε χώρα ανάλογα με το επίπεδο διαβίωση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε για να δούμε τι δυνατότητα έχουν πλέον τα κράτη-μέλη αφού του αφαιρούμε αυτά τα εργαλεία για να μπορούν ανεξάρτητα να αντιμετωπίζουν κρίσει. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το χάσμα στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών. Η Τραπεζική Ένωση δεν νοείται πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ολοκληρώσει το στόχο να φέρει πιο κοντά το επίπεδο διαβίωσης των κρατών μελών. Η τραπεζική κρίση στα κράτη-μέλη είναι κάτι που αφορά τις εθνικές ε, ε, κεντρικές τράπεζες και μόνο γιατί έχουν και την ιστορική εμπειρία να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους εθνικά προβλήματα. Βάλτσο, για ένα λεπτό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η Τραπεζική Ένωση είναι ένα μέσο μιας διαδικασίας ολοκλήρωσης που έχει ως στόχο να ε, αντιμετωπίσει ε, την κατάσταση, να προωθήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση χρησιμοποιώντας ως πρόπαση την τραπεζική κρίση και τη χρηματοπιστωτική κρίση. Ε, θυμάστε την επιστολή των πέντε προέδρων που λέει ότι θα πρέπει ο ΝΕ να ολοκληρωθεί και να εμβαθυνθεί. Προσωπικά πιστεύω ότι η, ε, είναι κάτι το ανέφικτο. Οι χώρες είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και η οικονομική τους ανάπτυξη δεν μπορούν να μπουν στο ίδιο τσουβάλι. Η ΟΝΕ, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, έχει χώρες ε, που είναι πιστωτές, άλλες χώρες που είναι ε, δανειολήπτριες και δεν λειτουργεί το μοντέλο. Η ενιαία Ευρώπη είναι αναποτελεσματική, δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή ηγεσία, έτσι κι αλλιώς ο κύριος Λάγκεν για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η παρούσα έκθεση είναι μια πολύ καλή δουλειά, επιμελής, με θετικά, μετά το πρώτο έτος της Τραπεζικής Ένωσης, αλλά δεν είναι αρκετά κριτικό το μάτι της ε, πρώτων. Ε, ο διαχωρισμός νομισματικής πολιτικής και εποπτείας των τραπεζών δεν είναι δεδομένος. Εδώ χρειάζεται τροποποίηση της συνθήκης και βλέπουμε που οδηγούμαστε. Ε, ε, έχουν αυξηθεί οι ποσοστό ιδίων κεφαλαίων σε όλη την Ευρώπη, αλλά οι χορηγήσει έχουν μειωθεί ιδιαίτερα στην Νότια Ευρώπη. Ε, δεύτερον, οι μεγάλες τράπεζες και οι μικρομεσαίες καλούνται να πληρούν τα ίδια κριτήρια. Από την αρχή δεν είχε προβλεφθεί έτσι, τώρα όμως εφαρμόζεται στην πράξη. Για ποιο λόγο και πού οδηγεί αυτή η γραφειοκρατία από 25.000 ευρώ και πάνω κάθε δάνειο θα πρέπει να δηλώνεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου αυτά τα πράγματα. Ε, και ε, ε, επίσης δεν λαμβάνεται ο κύριος Γκίγκολτ έχει βγάλει το αγαπημένο του θέμα ε, για τις ε, εγγυήσεις, για τα δάνεια, παρόλο που έχουμε αποφασίσει κάτι διαφορετικό. Και τέλος να θυμίσω πώς προέκυψε όλη αυτή η ιστορία. Η Τραπεζική Ένωση γεννήθηκε διότι η Ισπανία δεν ήθελε να μπει στο Ταμείο Διάσωσης. Γι' αυτή ε, την ευκαιρία έχουν χρησιμοποιήσει το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Γαλλία για να σώσουν την τράπεζα Ντέξια. Και θυμάμαι τον κύριο Αλμούνια που μέσα σε ένα 24ωρο ενέκρινε 24 ε, εκατομμύρια ευρώ ως εγγύηση για την δέξια μέσα σε 24 ώρες. Ο κύριος Μακάλιστε ζήτησε να σας κάνει ερώτηση. Μα είστε από την ίδια πολιτική ομάδα. Ε, αυτό είναι κατά ε, του πνεύματος της μπλε κάρτας. Η κυρία Μπερές, για 1,5 λεπτό παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να συμφωνήσω με τον κύριο Μπάλτ. Λέει πως ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε αυτά που αρχίσαμε. Διότι εάν δεν το κάνουμε, τότε, όπως λέγεται, κάνουμε αρκετά για να μας καταλογίζουν τι ευθύνε, αλλά δεν κάνουμε αρκετά για να μας αποδοθούν και τα εύσημα. Πρέπει λοιπόν να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια. Ε, Τι αυτή περιπτώσει μας λείπουν περισσότερα από αυτά που αναφέρατε. Θέλουμε backstop, αποθεματικό, ασφαλείας και χρειαζόμαστε εγγύηση καταθέσεων. Αλλιώς, ένα μας μπούμεραν θα στραφεί αυτό που καταφέραμε και θα πρέπει με αποφασιστικότητα αυτό το δρόμο να ακολουθήσουμε έχουμε φτιάξει όλη τη συζήτηση γύρω από την, ε, το θέμα της ε, μείωσης ε, των κινδύνων και του επιμερισμού τους. Πίσω από αυτή την υπέροχη έννοια όμως ε, ε υπάρχει μια άλλη ουσιαστικότατη συζήτηση που δεν γίνεται για, τα, για το εθνικό χρέος. Αυτοί οι υπέρμαχοι της διεθνούς προσέγγισης θέλουν ταυτόχρονα να μην λαμβάνονται υπόψη τα δημόσια χρέη με βιώσιμο τρόπο. Και ταυτόχρονα δεν θέλουν να ε, κερδοσκοπούν κάποιοι με τα δημόσια χρέη για να, ε, πώς, ε, με, το, τη μη υποβολή του στο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Μα δεν ε, είναι λογικό. Ευχαριστούμε. Ρόνεν Λέσνερ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά θα πρέπει να πληρώσουμε εμεί τα σασμένα για την Νότια Ευρώπη. είναι σίγουρο ότι εάν θεσπιστεί κάποιο τέτοιο κοινό σύστημα εγγύησεων στην ε, Ευρωζώνη. Εντάξει, το δεχτήκαμε αυτό στα πλαίσια τη έκθεση και εγώ συμφώνησα και βέβαια η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο για κάθε τραπεζική δραστηριότητα. Ε, γιατί ούτε ένα ευρώ δεν θα καταθέσει ε, κάποιος πολίτης εάν δεν έχει εμπιστοσύνη στην τράπεζα. Και οι τράπεζες και στον Βορρά διαφέρουν πάρα πολύ από ότι και οι τράπεζες στον Νότο. Επομένως ε, θα έχουμε αυτό το κοινό σύστημα το οποίο θα ασφαλίσει τις καταθέσεις σε βορρά και νότο και αυτό θα αυξήσει την εμπιστοσύνη προς το τραπεζικό σύστημα όλες τις Ευρώπης. Γι' αυτό και εγώ είμαι κατά της ε, έκθεσης Γκουαλτιέρη. Ευχαριστούμε κυρία Ματίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν μιλάτε για την, ε, το λογαριασμό που πρέπει να πληρώσουν οι νότιε χώρε, να ξέρετε ότι μεταφέρθηκαν χρήματα από τι νότιε χώρε στην κεντρική Ευρώπη για να σώσουν ε, την ε, τις εμπορικές τράπεζες της Γερμανίας πιο συγκεκριμένα καθώς και γενικότερα τις ευρωπαϊκές τράπεζες λεφτά διοχετεύθηκαν σε αυτές τις τράπεζες και δεν είναι το μόνο που χρειαζόμαστε. Πρέπει να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Δηλαδή, πέρα από το μάρκετινγκ δεν υπάρχει πολιτική και για την Τραπεζική Ένωση. Χρειαζόμαστε εγγύηση καθέσεων. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Από εκεί έπρεπε να αρχίσουμε. Ο ενίος μηχανισμός εξυγίανσης, ε, τι έχουμε να πούμε γι' αυτό, το ελάχιστο είναι ότι είναι μια ουτοπία και είναι ανεπαρκέστατος ο μηχανισμός. Ο, η ενιαία υποπτική αρχή, αυτό που άρχισε να ισχύει πρώτο, τι, ε, δεν ωφελεί σε τίποτα, διότι δύο χρόνια υπάρχει και όταν χρειάστηκε δεν λειτουργήσε. Αυτό συνέβη στην Πορτογαλία για την ε, ε, υποπτώχευση τράπεζα για δύο χρόνια έτσι. Όταν υπήρχε ο νέος εποπτικό μηχανισμός κανείς δεν την έλεγξε την τράπεζα, κανείς δεν μπορεί να τα εξηγήσει αυτά, κανένας ε, δεν επομίζεται τι ευθύνε. Είναι πραγματικά παραπληροφόρηση, κακό μάρκετινγκ. Ευχαριστούμε. Ντελάνια, ένα Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να πω στους συναδελφούς ότι χρειάζεται να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Και η Τραπεζική Ένωση είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της περασμένης θητείας. Αλλά δεν θα πρέπει ο πολίτης να αναλαμβάνει τις επιπολαιότητες και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι χρειάζονται τρεις πυλώνες. Ε, εποπτεία, εκαθάριση και εγγύηση καταθέσεων. Αλλά πολλά γίνανε σε εποχές κρίσης και ε, ε, ε, διακυβεύεται η αξιοπιστία των κρατών μελών και η εμπιστοσύνη. Τώρα υπάρχουν εθνικά συστήματα που εγγυώνται τις καταθέσεις. Δεν θα πρέπει να κάνουμε τώρα τόση φασαρία με τον τρίτο πυλώνα. Ενώ είναι κλονισμένη ακόμα η αξιοπιστία και μιλάμε για μείωση του ηθικού κινδύνου. Ας εφαρμόσουμε τις συμφωνίες για ε, τους δύο πρώτους πυλώνες, αλλιώς είναι χτίσματα στην άμμο αυτά που κάνουμε. Να αφήστε τον τρίτο πυλώνα, να ολοκληρώσουμε αυτά που συμφωνήσαμε και και όπως έχουμε και το κριτήριο no creditor wars, να έχουμε και το κριτήριο no member states wars. Και να μην χτίζουμε στην άμμο. Κυρία Ντελάγκε, ε, έχει μπλε κάρτα. Ο κύριος Μονό, τη δέχεστε παρακαλώ. Τη δέχεστε παρακαλώ. Κύριος Μονό. Ε, είμαι πολύ ευαίσθητος στα επιχειρήματά σας και τα καταλαβαίνω, αλλά σας ερωτώ το εξής. Ε, διαρκώς και ε, ε, να έως, μιλάτε για τους φορολογούμενους. Οι φορολογούμενοι δεν είναι καταθέτες. Ε, και δεν θέλουν ε, εγγύηση για τις καταθέσεις τους ή τις αποταμιεύσεις. Είδαμε τι έγινε στην Ιταλία το 2015 το Δεκέμβριο στις τράπεζες που επτόχευσαν. Δηλαδή για μένα φορολογούμενος ίσον πελάτης τραπεζών. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Ακριβώς. Και γι' αυτό κοιτάξτε τους κανόνες. Υπάρχουν κανόνες. Μέχρι 100.000 οι καταθέσεις είναι εγγυημένες από τα εθνικά συστήματα. Εάν τώρα οι τράπεζες είναι επιπόλαιες και δίνουν προϊόντα στους ε, πελάτες υψηλού κινδύνου χωρίς να τους ε, ενημερώσουν ότι είναι θέμα καταναλωτικό και όχι εγγύησης καταθέσεων, φοβούμε το εξή εγώ. Ότι αν τα κράτη-μέλη, και δεν κατονομάζω καμία χώρα, αλλά προσπαθήσουν να ε, αποφύγουν την αρχή του bail-in που έχει ως στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος και ο ηθικός κίνδυνος είναι σαν να λέμε ότι εντάξει δεν θέλουμε το bail-in αλλά ε, ε, μεταθέτουμε και μετακυλίουμε ε, το λογαριασμό στο φορολογούμενο άρα και στο κράτος. Και κάποια κράτη θέλουν να στείλουν το λογαριασμό σε ορισμένα άλλα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λέμε όχι Warsaw. Φερνάντες, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα, πρώτα συγχαρητήρια στον εισηγητή τον κύριο Γουαλτιέρη. Νομίζω ότι έχετε συνθετικά παρουσιάσει τις πρότασης των τελευταίων ετών για την οικοδόμηση αυτής της Τραπεζικής Ένωσης. Αυτό το, το, το, όραμα το τραπεζικό που πρώτα πρώτα αφορά τη σταθεροποίηση της οικονομίας με το ευρώ και μιλάμε για ανάμψη της οικονομίας οπότε και χρειάζεται για καλύτερη δημοσιονομική πολιτική πιο ρωμαλαία. Όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο όπως πάνε περισσότεροι συνάδελφοι και ε, μπράβο που υπάρχει όλη αυτή η πλειοψηφία για να προχωρήσουμε στον τρίτο πυλώνα. Αυτό χρειάζεται για την ασφάλεια των καταθέσεων και αυτό θα πρέπει να γίνει ταχαίως και θα πρέπει να γίνει πιο αποφασιστικά από το χρονοδιάγραμμα που έχουμε καταρτήσει εδώ στο Κοινοβούλιο και είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδου ε, αναθεώρηση από πλευρά νομική για το κρατικό χρέο. Θα πρέπει να περιορίσουμε του κινδύνου, θα πρέπει να υπάρχει μια εποπτεία και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια στους ολογισμούς των τραπεζών αλλά επίσης θα πρέπει να έχουμε και κάποια αλλαγή ποιοτική όσον αφορά το τι θα γίνει με το χρέος και έτσι να μπορέσουμε να ανασχέσουμε αυτή την κατάτμιση που υπάρχει στην Ευρωζώνη. Γιατί αυτό είναι το ζουμί, αυτός είναι ο σκοπός της Τραπεζικής Ένωσης. Οπότε εδώ υπάρχει μια αντίφαση και θα πρέπει να έχουμε μια κοινή αγορά από την μία μεριά αλλά από την άλλη μεριά έχουμε τις διαφορές και τη διαφορετική αντιμετώπιση των αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιώνας, υπάρχει μια ερώτηση από πλευράς του κυρίου Λάγκεν. Αποδέχεσαι την ερώτηση. Μάλιστα. Η ερώτηση. Συνάδελφε, είπατε ότι ήταν τεράστια επιτυχία, λέει η Τραπεζική Ένωση. Τώρα έχουμε τα προβλήματα ότι η νομισματική πολιτική και η εποπτεία των τραπεζών δεν είναι ε, διακριτά και η ΕΚΤ έρχεται και διαπιστώνει ότι είναι υψηλό ο κίνδυνος και θέλει να περιορίσει τα μετρητά που κυκλοφορούν το ένα και, θέλει να ε, καταργήσει τα, ε, το χαρτονομίσματα των 500 ευρώ. Εσείς το θεωρείτε αυτό επιτυχία ή το βλέπετε με κριτικό μάτι. Και θέλει να βάλει και αρνητικό επιτόκιο γιατί δεν παίρνει μπρος η οικονομία στην Νότια Ευρώπη. Όλα αυτά τα θεωρείτε θετικά εσείς. Ναι, ευχαριστώ. Εγώ νομίζω ότι να σωστή κατεύθυνση με την Τραπεζική Ένωση και τα προβλήματα που υπάρχουν για την Νομισματική Επιτροπή και για την Εποπτεία, αυτά νομίζω ότι υπάρχουν σε διάφορες χώρες όπω και στη δική μα. Και ε, αυτό συνεχίζεται γιατί άλλο είναι η νομισματική πολιτική και άλλο η εποπτεία. Οπότε τώρα έχουμε πρόβλημα για να μπορέσει να ανανύψει η Ευρωζώνη, αλλά αυτό το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με την νομισματική πολιτική. Το πρόβλημα είναι ότι ακριβώς δεν υπάρχει ένας ε, πυλώνας δημοσιονομικός και για το ότι κάποιες χώρες συνεχίζουν και έχουν πλεονάσματα πλεονάσματα τα οποία προκύπτουν στο, στο, στον, ε, στον προϋπολογισμό τους και αυτό προβληματίζει τις οικονομίες του Νότου. Κύριο Ζωκ, έχετε το λόγο και εσείς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Δεν έχω πολύ χρόνο. Οπότε απλώς θα σας πω δύο λόγια. Θεωρητικά το θέμα της εγγύησης των καταθέσεων από πλευράς Ευρωζώνης είναι μια συνέπεια που απορρέει λογικά από τα βασικά συστατικά της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Όμως υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις για το τι, πώς θα καλυφθούν ε, τα έξοδα αυτού του συστήματος. Μήπως θα τα πληρώσουν οι καταθέτες, οι πελάτες του συστήματος, γιατί στην ε, Πολωνία έχουμε ε, διάφορα αλλοδαπά κεφάλαια τα οποία έχουν επενδύσει στην αγορά και θεωρούν ε, αυτοί οι κύκλοι που έχουν επενδύσει ότι δεν είναι κάτι το θετικό αυτό το σύστημα παρά το ότι δεν ανήκουμε στην Τραπεζική Ένωση δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν εγγυήσει ότι οι δαπάνες του συστήματος πρόκειται να περιοριστούν γιατί θα υπάρξει κάποια άστοχη διαχείριση ή και πτώχευση τραπεζών σε άλλες χώρες. Κύριε Ντεμαζή, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απειλεί μια νέα οικονομική κρίση και χρηματοπιστική καζίνο αυξάνεται πιο γρήγορα από ε, την οικονομία και δεν ξέρουν οι σούπερ πλούσιοι που να βάλουν τα λεφτά τους. Και στην Ιταλία ε, ε, έχασε ο κόσμος τις οικονομίες μιας ζωής γιατί οι τράπεζες ήταν πόλες. Αυτή είναι η εποπτεία. Θα πρέπει να προστατεύονται οι μικροεπενδυτές, οι μικροκαταθέτες, όχι με παραθυράκια. Η ευθύνη των ε, μετόχων και των ε, καταθετών ε, θα πρέπει να είναι υπεύθυνη. Η Deutsche Bank κινδυνεύει ε, θα πρέπει η εποπτεία να διαχωριστεί από την νομισματική πολιτική για να μην μπορούν οι τράπεζες να συνεχίζουν να εκβιάζουν τους ε, φορολογουμένους. Χρειάζεται εγγύηση για τους μικροκαταθέτες και όχι για ε, εκείνους που τζογάρουν σαν να ήταν καζίνο. Και τα, τα μιευτήρια θα πρέπει να εξαιρούνται. Ευχαριστώ, Μάρκ. Πρόεδρε, Κάνουμε κάποια εκστρατεία για τον κατακαιρματισμό. Μπορείτε να λέτε «Α, μα, α, μας αρέσει η γραφειοκρατία, θέλουμε περισσότερο, όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα». Ε, σας βοηθάω για να κάνετε πιο αποτελεσματικά την εκστρατεία σας. θέλω να περάσουμε τώρα στη συζήτηση για τις τράπεζες. Και ευχαριστώ τον εισηγητή. Το βασικό πρόβλημα στην Ένωση δεν είναι η έλλειψη κανονιστικών ρυθμίσεων. Το αντίθετο ισχύει, διότι τώρα προσαρμοζόμαστε σε αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί και αρχίζουν να ισχύουν. Το αντίθετο είναι το πρόβλημα η έλλειψη των επενδύσεων, η έλλειψη ανάπτυξης. και προσπαθούμε να, να εμποδίσουμε τις τράπεζες από το να έχουν ρευστότητα και να ε, ε, τροφοδετούν τις αγορές. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί με καμία εργοδεσία δεν μπορούμε να αντισταθμίσουμε την έλλειψη ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης. Ας το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα διαχωρισμό ανάμεσα στα δύο είδη τραπεζών και πλειοψηφία δεν έχετε, οπότε δεν μπορείτε να το δείτε. Κύριε Χόκμα, γαλάζια κάρτα από, τον, ε, από την κυρία Φερέιρα, τη δέχεστε. Ναι. Κύριε Φεραίρα, ευχαριστώ κύριε Χόκμαν για τη δουλειά που έχετε κάνει για την BRRD. Θέλω να σας ρωτήσω ακριβώς για το χρέος. Ε, προϋποθέτεται ότι χρησιμοποιείτε το Μπέιλιν και άρα βαρύνονται οι καταθέτες. Θεωρείτε ε, ότι είναι βιώσιμο αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μιλάω για γερμανικές ε, τράπεζες, ε, διότι κρύβονται κάποιοι πίσω από τα ιδιωτικά κεφάλαια και το Μπέιλιν τελικά τους προστατεύει, δεν εφαρμόζεται σε αυτούς το Μπέιλιν και ε, κρύβονται πίσω από αυτό και θα ήθελα να ξέρω αν εσείς γνωρίζετε αυτή την κατάσταση και τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Απάντηση. Σας ευχαριστούμε κυρία Φερέιρα. Να σας πω το εξής. Ποιος είναι ο στόχος του Μπέιλιν. Ακριβώς οι καταθέτες να μην ε, πληρώνουν για τις ε, ζημιές, για τις απώλειες. Σε αυτή την ε, νομοθεσία BRRD και χαίρομαι που ήμουν συνυπεύθυνο μαζί σας εξάλλου για αυτό το ζήτημα αναζωογονήσαμε την χρηματοδότηση, την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών και σας ευχαριστώ. Στη Γερμανία, στη Σουηδία, στην Πορτογαλία αυτό τι σημαίνει, ότι δεν θα έχουμε χρήματα φορολογουμένων μέσα στον Μπελίν μέχρι να ασχοληθείτε και να λύσετε το πρόβλημα του 8%. Το πώς θα το κάνουμε εκεί μπορεί να δούμε διαφορές. Όλα τα κράτη-μέλη προσαρμόζονται τώρα στη νέα νομοθεσία. είναι σημαντικό αυτό να γίνει και στην Πορτογαλία και στην Ιταλία και στη Σουηδία. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαριάς, ένα λεπτό κύριε πρόεδρε ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός που συστάθηκε στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης για να συμβάλει δήθεν στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος αποδείχθηκε ότι δεν επαρκεί για την εξυγίανση των τραπεζών. λόγω της οικονομικής κρίσης εκατομμύρια ευρώ δημόσιου χρήματος διατέθηκαν για τη διάσωση των τραπεζών επιβαρύνοντας το δημόσιο χρέος των κρατών και όλα αυτά τη στιγμή που τα κεφάλαια που διατέθηκαν για την ανεργία είναι ελάχιστα στην ελλάδα έγιναν τρει ανακεφαλαιοποιήσει τραπεζών που αύξησαν το δημόσιο χρέο και κοινωνικοποίησαν τι ζημιέ των τραπεζών. μάλιστα με το τρίτο μνημόνιο πωλήθηκαν ξανά οι τράπεζε σε ιδιώτες και κοράκια και αντί πινακίου φακή με αποτέλεσμα το δημόσιο να ζημιωθεί κατά 30 δισεκατομμύρια ευρώ. και σαν να μην έφτανε αυτό οι τράπεζε αφού διασώθηκαν πολλούν πλέον τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια σε κερδοσκοπικά φαντ και κοράκια

ότι τώρα έχουμε μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση θα είναι καλύτερο και θα έχουμε πιο πολλές τράπεζες και πιο μεγάλες ε, και τι θα γίνει με τις μικρές τράπεζες στην ε, χώρα σας αυτές πρόκειται να τις ε, καταπιούν οι μεγάλες τράπεζες και έτσι να έχουμε κάποια, κάποιες τράπεζες τέρατα τι νομίζετε ότι προς τα εκεί πάμε θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση κυρία Μαριά η απάντησή σας στην Ελλάδα η λύση που δόθηκε για τις μικρές τράπεζες και ιδίως για τις μικρές στεγαστικές τράπεζες είναι απαράδεκτη. Και είναι απαράδεκτη διότι αρκετές από αυτές έπρεπε να έχουν στηριχθεί. Όμως δεν στηρίχτηκαν οι μικρές αυτές τράπεζες με αποτέλεσμα να, να μπουν σε εκαθάριση. Πιστεύω ότι πρέπει να στηριχθούν οι τράπεζες οι οποίες είναι στην περιφέρεια οι συνεταιριστικές τράπεζες διότι αυτές είναι που συμβάλλουν στην πραγματική οικονομία. σε σχέση με την διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης στην ελλάδα αυτό που είδαμε ήταν να ξαναπάρουν αντί πινακίου φακής οι ιδιώτες τις τράπεζες που είχαν πριν και έτσι το δημόσιο να χάσει 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ρομπέρτο Γκολτιέρη για την έκθεσή του, καθώς επίσης και εκείνους που συνεισέφεραν. Είναι εξαιρετική έκθεση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο κύριο Χιλ και ε, σύνολη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονός ότι επιτέλους έχουμε μια νομοθετική πρόταση που έχει να κάνει με τον τρίτο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης που είναι σίγουρα ε, ο πιο περίπλοκος στην επίτευξή του και το σύστημα και το μηχανισμό εγγύσεων των τραπεζικών καταθέσεων. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής κύριε Επίτροπε. Με έκπληξη άκουσα κάποιες δηλώσεις που έκαναν πρόεδροι σημαντικών ε, ευρωπαϊκών τραπεζών, οι οποίοι θεωρούν, διοικητές δηλαδή, ότι ε, δεν πρέπει να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια και ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης είχατε κι εσείς αρκετά προβλήματα. Νομίζω θα πρέπει να συνεχίσουμε να το συζητάμε με τους επικεφαλείς των τραπεζών, ε, να τους πείσουμε ότι είναι σημαντική η Τραπεζική Ένωση και παραμένει. Θέλω να σας πω κάτι που συμβαίνει στη χώρα μου. Οι τράπεζες έχουν βαρεθεί να πουλούν στο 10% τα κόκκινα δάνεια, στο 10% της ε, ανομιστικής τους αξίας και καμιά φορά ε, δεν μπορούν να δώσουν ε, δάνεια καθόλου. Ο κύριος Χένκελ στην αρχή Τραπεζική Ένωση είχε προβλεφθεί ως εποπτεία και όλοι σκεφτόμασταν ότι θα έπρεπε να συζητάμε για τις τράπεζες και να τις επεπτεύουμε και όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Στο μεταξύ Γερμανοί, συνταξιούχοι και καταθέτες έχουν καταλάβει ότι πρόκειται για την αμοιβεοποίηση και κοινοτικοποίηση του κινδύνου. Δηλαδή ε, ε, θα πρέπει ε, να έχει συνυπευθυνότητα ο Γερμανός καταθέτης για το τζογάρισμα κάποιων ανεύθυνων ξένων τραπεζών. Τι λέει η δική μου εμπειρία. Όταν όλοι είναι υπεύθυνοι για τα πάντα τότε ουδής είναι υπεύθυνο για τίποτα. Αυτή η Τραπεζική Ένωση με αυτόν τον τρόπο που έχει δημιουργηθεί είναι τελείως ανεύθυνη. Τσέτερουμ τσέντζιον έλεγαν οι Λατίνοι. Και εγώ πιστεύω ότι το ευρώ στην Ευρώπη οδηγεί μόνο σε διχόνοια και σε έρηδες και θα πρέπει να καταργηθεί. Ο κύριος Φέρμπερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Αν δούμε πώς έχει η κατάσταση σήμερα μια φωτογραφία της Τραπεζικής Ένωσης θα διαπιστώσουμε ότι η οδηγία καθάρισης των τραπεζών δεν έχει εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη ε, ούτε τα ισχύοντα για την εγγύηση των καταθέσεων και ταυτόχρονα ακούμε νέες προτάσεις και παρακαλώ πάρα πολύ να φροντίσουμε πρώτα να εφαρμόσουμε αυτό που ήδη έχουμε αποφασίσει ως κανονιστικό πλαίσιο σε όλα τα κράτη-μέλη και να εφαρμόζεται και να υλοποιείται σωστά πριν προχωρήσουμε σε νέες προτάσεις όπως είναι η τελείως λάθος πρόταση ε, ε, για το ΕΔΙΣ, για το κοινό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Στη συνέχεια, πού είναι η αρχή της αναλογικότητας. Όλα τα προβλήματα στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να λύνονται με ευρωπαϊκή εποπτεία. Παράδειγμα ε, ε, η συμμετοχή στο Ταμείο Καθάρισης ξαφνικά φέρνει προτάσεις σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι μεγάλες τράπεζες πρέπει να δίνουν λέει λιγότερα και οι μικρές περισσότερα. Ε, οδηγείς για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει 4 και για τις πιο μικρές επενδύσεις και το Anacredit που είναι αυτή η τράπεζα δεδομένου. Τι να τα κάνουμε όλα αυτά. Χρειάζεται πολλή δουλειά να εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε αποφασίσει πριν φέρνετε νέες προτάσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία, κυρία Χίμπνερ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Πρώτα ευχαριστώ η Τραπεζική ένας κατά τη γνώμη μου είναι το πιο πετυχημένο ευρωπαϊκό όραμα το οποίο ακολούθησε ε, την χρηματοοικονομική κρίση και έχουμε τώρα το bailout μετά από την παγκόσμια λύση του bail-in έχουμε μας τώρα τις νέες ανάγκες του συστήματος που, τις οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούμε αλλά ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί 100% η πρόκληση τώρα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία προς τους ε, επενδυτές και τους άλλους εμπλεκόμενους παράγοντες της ε, αγοράς και ε, ιδίως ε, θα πρέπει να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους και θα πρέπει να υπάρξει κατανόηση του τι υπέρ και τι κατάχει το Μπέιλιν. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι αποκλήσεις έχουμε όταν έχουμε ε, εφαρμογή του BRD γιατί βλέπουμε ότι οι πιστωτές θα πρέπει να λαμβάνουν τα χρήματά τους και έτσι θα υπάρξει προβληψιμότητα και αξιοπιστία στο σύστημα και θα έχουμε πιο θεμητές συνθήκε ανταγωνισμού και σε αυτό θα συμβάλλει περισσότερη εναρμόνιση. Ευχαριστούμε κυρία Χίμπνερ. Και τώρα έχουμε την διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Μαυρίδης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στον εισηγητή για αυτή τη σημαντική έκθεση και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι προτού εμπλακώ στην πολιτική κύριε πρόεδρε είχα ακούσει ότι στην ευρωπαϊκή ένωση έχουμε κοινού κανόνες αλλά πολλές φορές αυτοί οι κοινοί κανόνες δεν είναι αμερόληπτοι. και αυτό είναι που έχουμε μπροστά μας τώρα. όταν η τραπεζική ένωση σχεδιάστηκε εξ αρχής κύριε επίτροπε η τραπεζική ένωση είχε και θα έχει νόημα εφόσον θα περιλαμβάνει και τους τρεις πυλώνες και φυσικά την εγγύηση των καταθέσεων. θυμάμαι όταν διοριστήκατε και είχαμε αυτή τη συζήτηση χωρίς τον τρίτο πυλώνα η ένωση είναι όχι απλώς λειψή είναι μεροληπτική εναντίον μικρών τραπεζών και μικρών κρατών μελών. οι καταθέτες πρέπει να τη χάνουν τη ίδια μεταχείρισης που δεν τη χάνουν οι τράπεζε πρέπει να τη χάνουν των ίδιων ευκαιριών που δεν τη χάνουν γι' αυτό λοιπόν όσο καθυστερεί τόσο περισσότεροι οι κίνδυνοι ελοχεύουν. Ο κύριος Σβάμπ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, η Τραπεζική Ένωση είναι όντως μια δύσκολη δοκιμασία ενώπιόν μας. Και θα ήθελα να σας κάποιος προηγουμένως. Συνήθως στην πολιτική θα πρέπει να αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα. Η Ευρωζώνη είναι γεγονός. Οπότε αυτά που λένε οι συνάδελφοι συντηρητικών και μεταρρυθμιστών απέχουν ε, πόρο από την πραγματικότητα. Πρέπει να βρούμε λύση εντός της ε, ΟΝΕ. Ε, για ποιο λόγο έχουμε τράπεζες για να εξυπηρετούν την πραγματική οικονομία. Είδαμε σκάνδαλα στην τραπεζική κρίση και τα ξεχάσαμε αυτά. Σωστά δημιουργήσαμε πολλούς νέους κανόνες, αλλά παρακαλώ κύριε Επίτροπε, κοιτάξτε τι γίνεται η πραγματική οικονομία. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να βοηθάει χωρί γραφειοκρατία την πραγματική οικονομία, επαναλαμβάνω. Και ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεση αυτή και τι αντίστοιχε παραγράφου. Σα Ευχαριστώ πολύ. Διάκασε ένα λεπτό. Αυτή αυτή η Τραπεζική Ένωση δεν έχει λύσει κανένα πρόβλημα. Τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι τώρα είναι ανεπαρκή και αυτά για τις εξηγιάνσεις των τραπεζών κτλ. Και ο πολίτης είναι αυτός ο οποίος καταδικάζεται να πληρώσει για τα μόνιμα προβλήματα των λεγόμενων συστημικών τραπεζών δεν έχει γίνει μια ουσιαστική προσπάθεια για την ελάχιστη ε, για τη μείωση μάλλον του κόστους το οποίο καλείται να πληρώσει ο ε, φορολογούμενος. Δυστυχώς δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα λύση και δεν θα υπάρξει αν δεν υπάρξει δημόσιος έλεγχος των μεγάλων ευρωπαϊκών πιστοτικών ιδρυμάτων. Brian. Θέλω να πω τρία και σύντομα. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη, για την απασχόληση η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τον τραπεζικό τομέα και θα πρέπει να προσαρμόσουμε ε, την Τραπεζική Ένωση όπου χρειάζεται. Επίση, έχει δίκιο τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει αυτή την αναθεώρηση. Άρα θα πρέπει να σταθούμε ειλικρινεί και να παραδεχτούμε ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσει όπου χρειάζεται. Αλλά να μην γίνει με τρόπο ευκαιριακό, γιατί πρόκειται για πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Ήταν εντολή προ το προηγούμενο και την προηγούμενη θητεία. Αλλά άμα κάτι δεν αποδίδει, άμα κάτι δεν λειτουργεί, να το αλλάζουμε. Επίση, τελικά είναι το θέμα τη ε, συγκυρία ε, τη συγκυρία τη δανειακή Πάρα προ τράπεζε δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ε, ζήτηση και αυτό κυρίω συμβαίνει στην ε, Ευρωζώνη. Άρα θα πρέπει να, να χρησιμοποιήσουμε κάποια αποθεματικά. Χρειάζεται ο ε, διάσωση, χρειάζονται τα stress test, αλλά τελικά θα πρέπει οι τράπεζε να μπορέσουν να βοηθάνε για την οικονομική ανάπτυξη, Αλλιώ πρόοδο δεν βλέπουμε. Κύριε Φλάνναγκαν, είστε το τελευταίο να λάβει το λόγο για ένα λεπτό. Η κυρία Φλάνναγκαν. 500 ε, εκατομμύρια ήταν το κόστος της διάσωσης των μη στιγμικών τραπεζών και αυτό είναι το κληροδότημα προς την Ιρλανδία και τώρα με αυτούς τους πυλώνες κάνουμε κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει τότε που το 1999 θεσπίστηκε το ευρώ Πέρσι επίση ε, χάσαμε 2 δισεκατομμύρια και 1 εκατομμύριο το 2014, το 2011 και τελικά φτάνουμε στο σύνολο των 6 εκατομμυρίων. Δηλαδή πάμε στο ότι έχουμε 25 δι τα οποία τώρα και αυτά πρέπει να διασπαθιστούν. Μα τι κάνει το Συμβούλιο, τι κάνει η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα ούτω ώστε να υλοποιήσουν αναδρομικά αυτού του κανόνε, να σώσουν την Ελλαδία και τον λαό τη από ε, αυτού του είδου την ζημιά των των 31 δις είναι η πέμπτη φορά που το λέω και δεν παίρνω απάντηση. Μπορεί να με ακούσει ο κύριος Επίτροπος να σταματήσουν εκεί την ε, κουβεντούλα και να δείξει επιτέλους κάποιον σεβασμό για αυτούς που εξέλεξε ο κόσμος. Σταματήστε να ασχολείστε με τον καφέ και να παίζετε στο ίντερνετ. Τι πρόκειται να κάνετε ούτω ώστε αναδρομικά να εφαρμόσουν κανόνες να σώσετε την Ιρλανδία και να κάνετε κάτι με αυτά τα 31 δις. Μα ίσως για την Ευρώπη να μην είναι πολλά λεφτά, αλλά για μας είναι πάρα πολλά. Πεινάει κόσμος λόγω αυτής της ε, ζημιάς. Οπότε ακούστε και σεβαστείτε την εντολή τη δική μου και των υπολείπων εδώ. Σας ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Χίλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε για την συζήτηση που προηγήθηκε η οποία είχε πολλά θέματα. Κάποια από αυτά είχαν σχέση με την Τραπεζική Ένωση, λέει ο κ. Επίτροπος. Στην ερώτηση για το αν το ποτήρι είναι μισοάδιο ή μισογεμάτο, θα πρέπει να απαντήσουμε ότι έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο και στα πλαίσια των stress test και ε, διαπιστώνοντας ότι έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα ισχυρότερο ε, με καλύτερη κεφαλαιοποίηση ε, και σε πολύ καλύτερη κατάσταση, πιο ανθεκτικό από ό,τι στο παρελθόν. Το θέμα είναι ότι δεν θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ, πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια και οι προτάσεις που έχουμε κάνει και μέσω της ανακοίνωσής μας για την μείωση του κινδύνου. Νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να πάρουμε κάθε μέτρο το οποίο θα βελτιώσει τα ε, επίπεδα εμπιστοσύνης, τον δίκτυ μάλλον εμπιστοσύνης. Η προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε έχει συνεχιστεί, έχουμε ανηλυμένες πλέον υποχρεώσεις, έχει υπάρξει πρόοδος και στην εφαρμογή των μέτρων αυτών ε, στα πλαίσια των τακτικών συνεδριάσεων του ΕΚΟΦΗΝ η πρόοδος που διαπιστώνεται από τη μία συνεδρίαση στην άλλη είναι σημαντικό. Σε σχέση με το θέμα που έθεσε ο κύριος Γκουαλτιέρη για το δημόσιο χρέος. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε με την προσεκτική ε, τακτική την οποία ακολουθεί και αυτό στις προτάσεις του. Ε, η προσπάθεια την οποία θα κάνουμε είναι κάτι το οποίο βρίσκεται υποσυζήτηση ε, και στην Οικονομική ε, Επιτροπή και επίσης είναι κάτι το οποίο απασχολεί και την Επιτροπή της Βασιλείας. Ε, το λεγόμενο backstop έχει τεθεί και αυτό. Τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει σε μια στάση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα το 2024 και αυτό έχει συμπεριληφθεί στην ανακοίνωσή μας για τα μέτρα μείωσης κινδύνου. Μέχρι τώρα λοιπόν, σχετικά με τις σκιώδεις λεγόμενες τραπεζικές δραστηριότητες, να πω ότι ο κανονισμός για τη χρηματοδότηση ομολόγων έχει ε, τεθεί σε λειτουργία από πέρυσι το MIFID όπως ξέρετε θα παίξει και εδώ έναν σημαντικό ρόλο οι νομοθετικές ρυθμίσεις και νομίζω ότι θα προχωρήσουμε γρήγορα ε, και ε, στις ε, αγορές κεφαλαίων. Θα είμαστε προσεκτικοί για να ανοιχνεύσουμε εγκαίρως κινδύνους που θα μπορούσαν να έρθουν στην επιφάνεια στα πλαίσια του shadow banking. Σχετικά τώρα με ένα θέμα το οποίο θέσατε και από τις δύο πλευρές, το θέμα της αναλογικότητας. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις έχει η νομοθετική ρύθμιση την οποία μέχρι τώρα έχουμε εφαρμόσει. Δεν το κάνουμε αυτό για να αμφισβητήσουμε τις αποφάσεις τις οποίες έχουμε λάβει αλλά να διαπιστώσουμε εάν έχουν εφαρμοστεί οι αποφάσεις αυτές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε επιτέλους τα πιστοτικά τραπεζικά κεφάλαια να περάσουν στην πραγματική οικονομία. Απαιτείται λοιπόν να δούμε ε, τι αποδείξεις πλέον έχουμε ε, επίσης θα πρέπει να ισορροπήσουμε τα ε, μακροπρόθεσμα και τα βράχυπρόθεσμα προληπτικά μέτρα. Είμαι λοιπόν ευγνώμων προς τον κύριο Γκολτιέρη και τους Σκιώδης για την προσπάθεια την οποία έκαναν και ελπίζω ε, σύντομα να συζητήσουμε εκ νέου για να συζητήσουμε για μια ακόμη φορά την πρόοδο η οποία έχει υπάρξει στην προσπάθεια ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής έχει το λόγο, ο κύριος Γκουαλτιέρη, για να κλείσει τη συζήτηση. Έχετε το λόγο κύριε Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συζήτηση που προηγήθηκε έθεσε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το βασικό χαρακτηριστικό της έκθεσης αυτής ήταν η προσπάθεια λεπτομερούς ανάλυσης των διαφόρων ε, πλευρών, αν θέλετε, ε, αυτού του πρώτου χρόνου εφαρμογής των αποφάσεων, να δούμε τι λειτουργήσε καλά, τι λειτουργήσε λιγότερο καλά, έχουν υπάρξει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις όπως είπε ο Γκίγκολντ και θα θέλαμε να προσκαλέσουμε όλους τους εμπλεκομένους σε μια ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΚΟΝΑ έτσι ώστε να δοθούν πιο συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτηματικά μας. Ε, τα θέματα MBA, τα θέματα των ΣΡΕΠ, e η ανάγκη ε, να καλυφθούν οι ανάγκες των μικρομεσαίων είναι θέματα τα οποία είναι δύσκολο να συζητηθούν σε επίπεδο ολομέλειας, ενώ τίθενται άλλα θέματα για τον διαχωρισμό των τραπεζών, για το bail-in, για το bail-out και τα λοιπά, ε, ταιριάζουν περισσότερο στην ολομέλεια. Όλες όμως αυτές οι συζητήσεις δεν πρέπει να βασίζονται σε ιδεολογήματα, αλλά πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένα δεδομένα. Οι κανόνες πρέπει να γίνουν, να γίνουν σεβαστοί. Οι κανόνες όμως οι ίδιοι πρέπει να επιτρέπουν να λαμβάνονται μέτρα τα οποία να μην λειτουργούν αρνητικά στην ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τα πράγματα εξελίσσονται σχετικά με θετικό τρόπο. Στη Γερμανία σαν παράδειγμα δημιουργείται ένα ίδρυμα το οποίο θα μπορέσει να αποτρέπει τα bail-in και να αποζημιώνει τους κατόχους ομολόγων. Νομίζω ότι πρέπει τα μέσα που έχουμε να τα χρησιμοποιήσουμε με ευφυή τρόπο. Πρέπει επίσης να πούμε ότι δεν προβλέπεται πλέον καμία χρήση ε, ε, των ε, χρημάτων των φορολογουμένων. Η πρόεδρος διακόπτει τον κύριο Γκουαλτιέρη. Όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν και στα πλαίσια της Βασιλείας. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι.